Good afternoon, Καλησπέρα, συνάδελφοι. Να σας καλωσορίσω και πάλι. Πρώτου ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία από την Σομαλία που μας επισκέπτεται. Η αντιπροσωπεία επισκέπτεται στην Βρυκλέ, της Βρυξέλλες στην προσπάθειά της να πείσει για την αναγνώριση του Σομάλιλαντ επικεφαλής είναι ο κύριος Μοχάμετ Μπηγιόνης που συνοδεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αντιπρόσωπο στις Βρυξέλλες, τον κύριο Ντουχά σας ε, καλωσορίζω λοιπόν εκ μέρους της Επιτροπής μας, στη συνεδρία μας. Θα γίνει συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το πώς οι δικές τους παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και βεβαίως σας καλούμε να παραμείνετε εδώ και στην ε, πορεία των εργασιών σας εδώ στις Βρυξέλλες θα χαρούμε πολύ να συναντηθούμε μαζί σας και να μιλήσουμε μαζί σας. Έχετε το ελεύθερο λοιπόν να μείνετε εδώ ή να ακολουθήσετε το δικό σας πρόγραμμα. Πάμε στο σημείο 8 λοιπόν της σημερινής διάταξής μας που είναι οι κύριες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στήριξη στο 11ο ΕΤΑ κονδύλιο χρηματοδότησης με αντίκτυπο. Θα γίνει ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Πιμ Βαν Μπάλεκομ, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Γνωρίζουμε ότι η ΕΤΕΠ έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στις χώρες ACP και έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια στο Impact Financing Envelope τον μηχανισμό που χρηματοδοτεί ιδιαίτερα ευάλωτες χώρες και υποστηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γυναίκες και νέους. Θα γίνει συζήτηση λοιπόν στην ε, Επιτροπή μας για το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σήμερα το πρωί είχαμε συζήτηση με τον ΟΑΣΕ, με τον ε, κύριο Σόχαϊμ. Τρεις εκθέσεις δικές μας σχετίζονται με τις δικές σας εργασίες. Η πρώτη αφορά την ε, χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η δεύτερη αφορά τους ε, πόρους στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες και η τρίτη αφορά τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά αφορούν και τις δικές σας εργασίες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πολλά μέλη της Επιτροπής μας είναι νέα μέλη και του Κοινοβουλίου, οπότε μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια, αν θέλετε, για το ιστορικό, για το υπόβαθρο της, ε, του οργανισμού σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και που με κάλεσατε στην Επιτροπή σας. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Όπως είπαμε, αντιπρόεδρος, υπεύθυνο και αρμόδιος για ζητήματα χρηματοδότηση και δανεισμού πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο συγκεκριμένα ACP, OCT, Νότια Αφρική και Τουρκία. Και οι υπόλοιποι φάκελοι αφορούν αρμοδιότητα των συναδέλφων μου. Όμως ε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτές τις επενδύσεις εν είδη σύντομη εισαγωγή. και βεβαίως να συζητήσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και να απαντήσω αν έχετε και εσείς ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είμαστε η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μοναδικό χρηματοδοτικό χρηματοπιστωτικό ε, ίδρυμα που δεσμεύεται να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, θεσπιστήκαμε υπό την συνθήκη της Ρώμης και ανήκουμε στα 28 κράτη-μέλη. 28 Υπουργοί Οικονομικών δηλαδή είναι η μετοχή μας. Είμαστε επίσης ε, ο μεγαλύτερος υπερεθνικός ε, δανειστής ε, στον κόσμο με όγκους δανεισμού έως και 70 δις ευρώ το χρόνο. Πέρσι το 2014 αγγίξαμε και τα 76 δις. Περίπου 90% του όγκου μα αφορά την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 7 με 8 δις ευρώ παρόλα αυτά, κατευθύνονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό το ποσό αυτό. Και κάνουμε αυτές τις επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Στις καθημερινές μας εργασίες ε, συνεργαζόμαστε από κοινού με την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία Δράσης και βεβαίως και με ευρωβουλευτές Θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και στην νέα κοινοβουλευτική θητεία, προκειμένου να στηρίξουμε με καλύτερο τρόπο τις εξωτερικές ε, πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕΠ λοιπόν είναι μια τράπεζα επενδύσεων με ε, σκοπό την ανάπτυξη, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως χρηματοδοτικό ίδρυμα στηρίζουμε οικονομικά βιώσιμα και τεχνικά εύρωστα έργα που πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια που θέτουμε και συνάδουν με όλες τις νομοθετικές ε, διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζονται από το Κοινοβούλιο αυτό. Στις επιχειρήσεις μας ε, εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από, τους, τις χώρες εταίρους για να προσδιορίσουν έργα με σημαντικό αντίκτυπο ως προς την ανάπτυξη. Εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από το επενδυτικό κλίμα ε, και περιβάλλον στην ε, περιφέρεια ή χώρα όπου λειτουργούμε. Στη διαχείριση λοιπόν, κράτος δικαίου είναι σημαντικά στοιχεία για μας για να βρούμε αξιόπιστους και ενδιαφέροντες εταίρους. Γιατί να θυμάστε ότι πάντα χρησιμοποιούμε σε ένα ποσοστό 30-50% μιας επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να χρηματοδοτήσουν από κοινού. Και αν υπάρχει χρηστή διαχείριση, κράτος δικαίου και ένα ευνοϊκό ε, επενδυτικό κλίμα, αυτό μας ευκολύνει και εμάς. παρότι είμαστε το μεγαλύτερο δημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον κόσμο, είμαστε μάλλον ε, μικρό ίδρυμα από την άλλη ε, με έδρα το Kingsberg στο Λουξεμβούργο, δεν εκπροσωπούμεθα λοιπόν παντού και έτσι υπάρχει σημαντική εξάρτηση ε, με τους εταίρους μας, όπως η Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων, η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και ε, στις διμερείς μας ε, σχέσεις όπως το KFW, AFD κλπ. Στηρίζουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και έτσι μειώνουμε αποτελεσματικά την ε, ανέχεια. Μετράμε τα αποτελέσματά μας από τα έργα μας και με χρηματοπιστωτικούς και μη όρους μέσω του λεγόμενου πλαισίου μέτρησης αποτελεσμάτων. Κάτι το οποίο ε, συστάθηκε πριν από δύο χρόνια, το 2012. Θέτουμε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη και οι προκλήσεις που συνδέονται με αυτήν στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τον ε, δημόσιο τομέα. Και ο ιδιωτικό ε, τομέα λοιπόν και η ανάπτυξή του είναι πολύ σημαντική και αυτό συνάδει και με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Αλλαγή. Η συμβολή της επιχειρηματικότητας ε, στην ανάπτυξη και τη μείωση της ε, ανέχειας αναγνωρίζεται και από την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Και ξέρω ότι και ένα από τα μέλη σας ασχολείται ιδιαίτερα με ζητήματα ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Τα συζητήσαμε και χθε μαζί του. Αλλά τώρα διαβάζει τα έγγραφά του, βλέπω. Όπως ξέρετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κινητήριες δυνάμεις ε, της οικονομίας και εντοπίζουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση προ τη χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Διοχετεύουμε πόρου προ ε, τι τοπικέ επιχειρήσει και τα αμοιβαία κεφάλαια και έτσι παρέχουμε χρηματοδότηση και σε μικρομεσαίε επιχειρήσει και σε μικροεπιχειρήσει και αναπτύσσουμε τοπικέ χρηματαγορέ. Αυτό ε, δημιουργεί με τη σειρά του ε, θέσει απασχόλησης, ανάπτυξη, συμβάλλει στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη ε, και σε μια κοινωνία και οικονομία χωρίς αποκλεισμού. Αν διαβάσετε και τις προβλέψεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για το 2015 σε αφορά την απασχόληση, η απασχόληση των νέων και πιο συγκεκριμένα των νέων γυναικών επιδεινώνεται. Παρά τα αποτελεσματικά στοιχεία προ την ανάπτυξη σε κάποιες ε, αναπτυσσόμενε χώρες. Στην Νότια Αφρική, για παράδειγμα. Γι' αυτό θέλουμε και εμείς να αυξήσουμε τι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Υλοποιήσαμε, για παράδειγμα, ένα περιφερειακό project στην Αφρική. Ε, σε συνεργασία με τοπικέ τράπεζες. Αυτό το project χρηματοδοτεί πιο ρηψοκίνδυνα έργα από μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, με ε, δάνεια ακόμα και 10 ετών. Με αυτό το μηχανισμό ε, δώσαμε χρηματοδότηση σε τοπικό νόμισμα και έτσι αντιμετωπίσαμε το ζήτημα των ε, μεταβλητών συναλλαγματικών συστημιών Και αυτό οδήγησε σε πολλά υποδάνεια προ τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον κοινωνικό και στον τομέα της υγείας και έτσι δημιουργήσαν πολλές θέσεις απασχόλησης στην τοπική οικονομία. Αλλά εμεί είμαστε και μια τράπεζα υποδομών ε, αρχικά Όλοι λένε ότι ασχολούμαστε μόνο με τα μεγάλα ψάρια, αλλά όταν μιλάμε και για μικροεπιχειρήσεις, ε, ακόμα και τις τάξεις των 2.000 Αμερικανικών δολαρίων. Προσπαθούμε πραγματικά λοιπόν να στηρίξουμε την ε, τοπική οικονομία, τον ε, κάθε μικρό καταστηματάρχη. Όμως ε, για την επιχειρηματικότητα χρειαζόμαστε και τις κατάλληλες υποδομές. Υπάρχει λοιπόν μία μικρή μετατόπιση προς τις μικροσύνε επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων μας αφορά τις υποδομές. Και έτσι έχουμε ε, ειδικά έργα για τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, του ύδατος ε, και του καθεξής. Με όλους τους τομείς χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει μέσω της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης και λαμβάνουμε και την ε, κλιματική αλλαγή υπόψη. Ε, προωθούμε τις ε, ενεργειακά αποδοτικές ε, μεταφορές και υποδομές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εξάγουμε λοιπόν την γνώση μας μέσω των εταίρων μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεντρωνόμαστε και στη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων Και πάλι η δράση μας είναι συγκρίσιμη με τα όσα κάνουμε στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι έως 50% είναι η χρηματοδότησή μας σε σχέση με το συνολικό κόστος του έργου. Και κινητοποιούμε περαιτέρω επενδύσεις από άλλους ε, θεσμούς, από άλλα θεσμικά όργανα, ε, φορείς δημόσιους ιδιωτικού για να ξεκινήσουν και να δρομολογηθούν αυτά τα έργα. Η τεχνική συνδρομή μας διευκολύνει την προετοιμασία και εφαρμογή των ε, έργων. Η τεχνογνωσία μας ε, και το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο που δίνουμε σε σχέση με τον εμπορικό κλάδο είναι ε, πλεονεκτήματα. Και αυτά τα πλεονεκτήματα δεν, ε, τα, δεν χαίρουν ιδιαίτερη εκτίμηση. Μάλλον, συγγνώμη, χαίρουν ιδιαίτερη εκτίμηση και μάλιστα πολύ σημαντικά θεωρούνται πιο σημαντικά από τις ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρουμε. Ελπίζουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο να μην αλλάξει, γιατί ακριβώς επειδή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί οι όροι μας, προσπαθούμε να τους ε, ε, μετακυλήσουμε προς ε, τον τελικό χρήστη. Ε, επίσης μπορούμε να κοινοτοποιήσουμε και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και να τα αναμίξουμε με τους δικούς μας πόρους και ιδιαίτερα για χώρες ε, χαμηλών εισοδημάτων βοηθάμε να διασφαλίσουμε ότι συνάδουν οι όροι μας και με την βιωσιμότητα του χρέους. Είναι ένα από τα στοιχεία του ε, σχεδίου Juncker, μια μετατόπιση από τις καθαρές επιδοτήσεις προς την ε, ανάμειξη των δύο διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης και εγγυήσεων κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. και έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση και πολλοί στηρίζουν ε, αυτές τις ε, αναπτυξιακές ε, πολιτικές. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της αυτή τη μορφή χρηματοδότηση είναι το ελληνικό πάρκο στην λίμνη Τουρκάνα με 310 ΜΒ ικανότητα σήμερα είναι ε, το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη τέτοια επένδυση στην ιστορία της ε, Κένιας και το συνολικό κόστος είναι 625 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς ε, δανείζουμε 200 εκατομμύρια ευρώ, ακόμα 25 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό, Ευρωαφρικανικό Τρασάντι Υποδομών που επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις επενδύσεις στις περιφερειακές υποδομές και σε έργα βιώσιμης ενέργειας στην υποσαχάρια Αφρική. Και έτσι μαζί με τις επιδοτήσεις και τον δανεισμό των Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιτρέπουμε να αρχίσουν έτσι οι εργασίες που θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2017. Θα ολοκληρωθούν μάλλον το 2017. Δεν θα τα πω όλα γιατί θα ήθελα να στραφώ σε κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό από ανθρωπιστική σκοπιά. σκοπιά. Ε, η κρίση του ιού έμπολα στην Δυτική ε, Αφρική. Η ΕΤΕΠ δεν ε, είναι ανθρωπιστικό ίδρυμα που παρέχει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Ε, στο διεθνές πλαίσιο υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που είναι πλέον κατάλληλοι όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ούτω καθεξής. Όμως ως Ευρωπαϊκή Τράπεζα και εμείς ε, ασχολούμαστε με αυτή την ε, περιοχή και συνεχίζουμε να λειτουργούμε εκεί. Στα τέλη του 2014 δώσαμε δάνειο 60 εκατομμύριων ευρώ για να αναβαθμίσουμε υδροελεκτρικές εγκαταστάσεις στη Γουινέα και έτσι δώσαμε καθαρή ενέργεια σε περισσότερους ανθρώπους. Έτσι και με, είναι και με ευνοϊκού όρου για να έχει αυτή η χώρα. Μετά, τον Οκτώβριο συγχρηματοδοτήσαμε σημαντική αναβάθμιση του ε, διεθνού αερολιμένα Ρόμπερτ στη Μονορόβια της Λιβερίας. 50 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων πήγαν στην Bavaria Nordic για ε, να ε, επιταχύνουμε τις διαδικασίες ανάπτυξης ενός ε, εμβολίου κατά του έμπολα. Σε ένα project διασύνδεσης 75 εκατομμύριων ευρώ, ακτή του Ελεφαντοστού, Λιβερία, Σιέρα Λεώνη και Ουινέα. Πολύ σημαντικό αυτό το έργο για την οικονομική ανάπτυξη δεν καθυστερεί παρά τα προβλήματα και υπό εξέταση είναι ένα project ε, διανομής ε, ύδατος στο Μάλι, το αντίστοιχο project υποδομών στη Σήμαντου στη Γουινέα και ε, μικροχρηματοδοτικά έργα στην περιφέρεια. Επομένως μπορούμε συνοπτικά να πούμε ότι εξακολουθούμε να ασχολούμαστε ιδιαίτερα ε, και με μεγάλη αφοσίωση σε αυτή την ε, περιφέρεια, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την ε, Κομισιόν, τον ΠΟΗ και άλλα θεσμικά όργανα. Προσπαθούμε διαρκώς να αυξάνουμε την προστιθέμενη αξία των έργων που χρηματοδοτούμε μέσω του συνδυασμού και της ικανότητας μας να επεκτείνουμε τα εργαλεία όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου και τις, τις ικανότητές μας προσπαθούμε πάντοτε να ε, καταλήγουμε και να φτάνουμε σε νέους δικαιούχους και να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο που έχουμε ως προς την ανάπτυξη. Και όπως είπαμε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με, το, ε, με τα 500 εκατομμύρια ευρώ του IFE που συμφωνήθηκαν ε, την προηγούμενη χρονιά που μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε έργα με υψηλότερο κίνδυνο. Οι τομεί εστίασή μα είναι οι κοινωνικές και δημογραφικές ε, προκλήσεις, η απασχόληση των γυναικών, η επιστημιστική ασφάλεια και η ανάκαμψη έπειτα από περίοδο συγκρούσεων. Την τελευταία χρονιά έχουμε ήδη εγκρίνει τρία project. Το project Novastar, ένα ταμείο για αφρικανικές επιχειρήσεις σε πρώιμο στάδιο, με στόχο την... Ε, ε, την χρηματοδότηση αγορών ε, και πολιτών με χαμηλό εισόδημα, κάτι που θα επιτρέψει στους ανθρώπους αυτούς να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμο, τρόφιμα νερά, νερό και υγεία. Επίσης, ε, χρηματοδοτούμε, κάνουμε επένδυση στο TCX, σημαντικό έργο για μικρές και μισές επιχειρήσεις. Και τέλος, με την συμμετοχή μας στο ε, χρηματοδοτικό μηχανισμό Καραϊβικής και ε, Ειρηνικού προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και αναμένουμε ότι, ότι τουλάχιστον 128.000 δικαιούχοι θα είναι γυναίκες. Το 2015 θα είναι η χρονιά όπου θα υιοθετηθούν οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα διαμορφώσουν ε, με τη σειρά τους τη δική μας ατζέντα για την ανάπτυξη. Η καταπολέμηση της ε, ανέχειας και η ενίσχυση της ευημερία παραμένουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, όμως και οι νέοι αυτοί στόχοι θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ε, διαχειριζόμαστε ζητήματα όπως είναι η χρηματοδότηση, ενέργεια, τεχνολογία και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στις παγκόσμιες προσπάθειες που καταβάλλονται μέσω απτών ε, έργων που χρηματοδοτούμε και προσπαθούμε να διαδραματίσουμε από την πλευρά μας το δικό μας ρόλο όσον αφορά την ε, συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιώσιμη ανάπτυξη μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο που έχουν τα έργα που χρηματοδοτούμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο, την Κομισιόν και βεβαίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση και για ε, ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε να μου θέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, συνάδελφοι. Ο κύριος Νόιζερ πρώτος και μετά η κυρία Ραφέρα Μπαστερέτσι. Ευχαριστώ κύριε Κομ για την παρουσία σας. Νομίζω στα βασικά σημεία του έργου σας συμφωνούμε ιδιωτικέ επενδύσεις. Παρά το γεγονό ότι κάθομαι στην αριστερή πλευρά της αίθουσα. νομίζω ότι στην Ολομέλεια την χάνουν τη ε, έγκριση της πλειοψηφίας. Μια ερώτηση. Τέσσερις φορές το χρόνο συζητούμε με συναδέλφους από τις αφρικανικές χώρες. Και μας θέτουν το ερώτημα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν συγκεκριμένα τα κονδύλια τα, ε, και η χρηματοδότηση. Η δική σας συμβολή ποια είναι στην πρακτική υλοποίηση ενός έργου όταν ένα κοινοβούλιο ή μια κυβέρνηση κάποιας χώρας λέει ότι θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις για παράδειγμα στην ανανεώσιμη, ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι συμβαίνει, εκεί παρεμβαίνετε εσείς, περιμένετε πρώτα να ε, ε, κάνει κάποιες κινήσεις η Κομισιόν, το κάνετε μαζί, υπάρχει κάποιος συντονισμός, μήπως μπορείτε να μας ε, πείτε ορισμένα στοιχεία, ώστε και εμείς να έχουμε κάτι να απαντούμε στους συναδέλφους. Και η άλλη ερώτησή μου αφορά ε, γενικά τις επενδύσεις. Το 90% είπατε ότι των επενδύσεων γίνονται στην ε, Ευρώπη, 10% κατευθύνεται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει κάποια τάση από τη δική σας πλευρά να αυξηθεί ο όγκος ε, της χρηματοδότησης που κατευθύνεται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόεδρος. Θα μαζεύουμε δύο-τρεις ε, ερωτήσεις γιατί έχουμε χρόνο. Η επόμενη ε, μιλήτρια είναι η κυρία Δαθέρα Δαστερέτσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε κύριε Βαμβάλεκομ για την παρουσίασή σας. Και για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Μ' ακούτε? Δεν ξέρω αν έχετε βρει το σωστό κανάλι. Εντάξει, ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και την παρουσία σα εδώ σήμερα στην Επιτροπή Ανατοχιακών Υποθέσεων και που σκεγγραφίσατε τις βασικές αξίες ε, που διέπουν το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων. Σα θεωρούμε καλό εταίρο μα, ιδίω ε, σε μία δύσκολη εποχή, όπου δύσκολα μπορεί κανείς ε, να διασφαλίσει αυτό το τριπλό α που είναι εξαιρετική βαθμολογία. Κάτι το οποίο θα ήθελα να δείξω που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την εικόνα της ΕΤΕΠ. Μιλώσετε για βιώσιμα έργα που είναι τεχνικά βιώσιμα λοιπόν και εφικτά και ε, συνάδουν και με τις ε, ανάγκες των ελλογοχωρών Συμφωνώ ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την προσθέμενη αξία των χρηματοδοτούμενων έργων. Θα ήθελα να αναφερθώ ένα συγκεκριμένο έργο στη χώρα μου, την Ισπανία το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την ε, τράπεζά σας. Αφορά ένα σχολείο στην ε, Βαλένθια, όπου για πολλά χρόνια οι μαθητές έκαναν ε, μάθημα σε προκάτ αίθουσες, το οποίο βεβαίως δεν είναι κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Τώρα η ΕΤΕΠ παρήχε μια οικονομική χρηματοδότηση, όμως δεν ολοκληρώθηκε το έργο, πέρασαν τα χρόνια, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το έργο, δεν εντάσσεται στην πρόταση που ενέκρινε η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτή την υπόθεση, γιατί εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα για ένα τέτοιο είδος έργου που υλοποιείται σε ένα κρατός μέλος. γιατί ήταν σημαντικό το ποσό, 800.000 ευρώ λοιπόν. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί οι μαθητές ακόμα σε αυτές τις προκάτ κάνουν μάθημα. Η Επιτροπή είπε ότι αναλύατε το σχέδιο δράσης, η τοπική αυτοδιοίκηση της Βαλένθια είπε ότι θα το εξετάσει, δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Εσείς θεωρείτε ότι έχει ευθύνη η ε, τοπική κυβέρνηση της Βαλένθια για το έργο υποδομών ως εκπρόσωπος των πολιτών της Ισπανίας θα έλεγα ότι εμείς στηρίζουμε την αξία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για να στη διασφάλιση ε, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το συγκεκριμένο έργο. Επόμενος ο ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Πράγματι συναντηθήκαμε το πρωί πολύ ευχαριστά, χθε μάλλον, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς ενθαρρύνεται μερικές αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τον τομέα των υπηρεσιών χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από όλη τη φάση των εθνικοποιήσεων που χρειαζόταν μέχρι τώρα, να προχωρήσουν δηλαδή. Βέβαια χωρίς εξηλεκτρισμό δεν γίνεται τίποτα. Με τον εξηλεκτρισμό όλα γίνονται δυνατά. Χρηματοδοτείται αρκετά έργα εξηλεκτρισμού ως εταίροι ώστε σε μια πρώτη φάση να παραχθεί ο εκτισμός και μετά ίσως να απολυθεί σε δίκτυα στην κυβέρνηση κτλ. Ξέρω ότι η Διεθνή Βαγκόσμια Παγκόσμια Τράπεζα δεν συμβάλλει και πολύ σε τέτοια έργα. Μήπως εσείς μπορούσατε να συμπληρώσετε υδροηλεκτρικά έργα. Τι χρηματοδοτούμε ακριβώς δηλαδή από τα βασικά, τις βασικές υποδομές. Ίσως τρεις-τρεις ερωτήσεις για να μην είναι πολλές μαζί. Πρώτον του κυρίου Νόιζερ. Δώστε μου κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τι είναι κύκλος έργου. Στην αρχή συζητάμε με τους εταίρους μας το πρόγραμμα και μετά και με σας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τα επόμενα συνήθως 7 χρόνια. Έχουμε και την εξωτερική εντολή δανεισμού και πρέπει να καθορίσουμε τι θα συμφωνηθεί μεταξύ των ενωσιακών εταίρων και των οργάνων. Τους στόχους αυτούς προσπαθούμε να δούμε αν συνδυάζονται με τους στόχους των χωρών όπου επενδύουμε και μας ερωτήσατε και χθες, μας ερωτήθηκε και χθες πώς επιλέγονται τα, τα προγράμματα, τα έργα. Όπως σας είπα εμείς είμαστε αναπτυξιακή τράπεζα σημαντικός παράγων, ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο περίπου επενδύουμε στις χώρες ΑΚΕ και στη Νότια Αφρική 1,1 δις σε άλλες χώρες και είμαστε πολύ σημαντικοί παίκτες διεθνώς. Η Παγκόσμια Τράπεζα μας συζητάει πολλές φορές και η ISU αν, μας ρωτάει αν ενδιαφερόμαστε να συμβάλλουμε σε ορισμένα έργα και προγράμματα. Το μελετούμε και μετά λέμε ναι ή όχι. Αφού υπογραφεί ένα σχέδιο ή πρόγραμμα ή έργο, ερχόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση της ενδιαφερόμενης χώρας για να δούμε αν συνδυάζεται και με άλλα. Αυτό είναι ο πιο φυσικός τρόπος νομίζω λειτουργίας μας. Εξάλλου πρέπει να εγκριθεί κάθε μια από τις επενδύσεις και από τη χώρα, την ενδιαφερόμενη χώρα. Μπορεί να υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης που δεν, δεν την ενδιαφέρουν. Κάτι συνεννοούμαστε και με την Κομισιόν. Νομίζω είναι πολύ φυσική διαδικασία. Τώρα για το 10% και το 90%. Επιτρέψτε μου να σας πω ειλικρινά ότι είναι λίγο τεχνητό αυτό το θέμα έτσι όπως παρουσιάζεται. Με το σχέδιο Juncker και την αύξηση των κεφαλαίων μας οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θέλουν τώρα να δώσουν έμφαση στις επενδύσεις μέσα στην Ευρώπη αλλά ειλικρινά σας λέω ότι οι αναδυόμενες αγορές εκτός της Ένωσης είναι κάτι που μας ενδιαφέρει επίσης και είναι κάτι που θα βοηθήσει και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν παρουσία στην Αφρική. Δεν είναι ένα πράγμα ασπρόμαυρα. Και μάλλον δεν έχει έρθει ακόμα επομένως η ώρα να τα αναθεωρήσουμε όλα αλλά ο διαχωρισμός μεταξύ δανειοδότησης εντός και εκτός της Ένωσης σε λίγο δεν θα υπάρχει η διάκριση. Θα γίνουν αυτοί, αυτά τα δύο είδη δανειοδότηση συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και Εμείς έχουμε ήδη αρχίσει να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ δανειοδότησης μέσα και εκτός ένωσης. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Τρίτο θέμα. Είπα 7 δισεκατομμύρια εκτός της Ένωσης χρηματοδοτούμε, 1 δισεκατομμύριο στις χώρες ε, και κτλ όπως σας τα είχα κατανείμει οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες της πολιτικής γειτονίας φυσικά έχουν προτεραιότητα. Αυτό πρέπει να τα δείτε όπως κατανέμονται. Για εκείνο το σχολείο στη Βαλένθια τώρα. Μας ρωτάνε πολύ ποιος σας ελέγχει, ποιος σας... Εμάς μας ελέγχουν 28 κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό. Επίσης η Γόλαφ, η Κομπισιόν και έχουμε και δικούς μας μηχανισμούς ελέγχου δημοσιονομικών ελέγχων κτλ. για την εποπτεία. Τώρα τι έγινε με τη Βαλένθια δεν ξέρω τι πήγε στραβά δεν είμαι υπεύθυνο για κάθε επιχείρηση και ειδικά στην Ισπανία. Θα ρωτήσω Ισπανούς μου συναδέλφους και θα επανέλθω με πιο συγκεκριμένη απάντηση. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Να είστε βέβαιοι πάντως ότι θα έχετε απάντηση στο ερώτημά σας. Κανονικά δεν χρηματοδοτούμε ένα μεμονωμένο σχολείο. Τις περισσότερες φορές έχουμε ένα γενικό επενδυτικό πρόγραμμα ας πούμε για την περιοχή της Βαλένθια που μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκατοντάδες σχολείων με ύψος μέχρι και 100 εκατομμύρια και όλα αυτά δεν δίνονται με μιας αλλά υπάρχουν φάσεις του έργου δεν ξέρω σε ποιο και ποια χρονική στιγμή του προγράμματος κάτι πήγε στραβά. Και γι' αυτό σταμάτησε μάλλον το πρόγραμμα. Θα επανέλθω πάντως αφού πληροφορηθώ από τον Ισπανό συναδελφό μου ή θα σας τα πει ο ίδιος. Βέβαια υπάρχει μετατόπιση από τις υποδομές στη μικροχρηματοδότηση γιατί η κατάσταση με την ανεργία στην υποσαχάρια Αφρική είναι πολύ σοβαρή και αυτό αγνωρίζεται και από όλους μας τους εταίρους αλλά είναι αδύνατο να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς τις κατάλληλες υποδομές όπως είπατε τον εξηλεκτρισμό. 80% των κατοίκων της Μουσαχάριας Αφρικής δεν έχουν πρόσβαση στον εξηλεκτρισμό ή στον ηλεκτρισμό. Και αυτή είναι μια από τις προτεραιότητες μας ώστε να υπάρξει τουλάχιστον μια αρχή οικονομικής ανάπτυξης υποδομές. Υπάρχει ένα πολύ επιτυχημένο αφρικανικό καταπίστευμα ή trust fund για υποδομές και επενδύουμε και σε ηλεκτροδοτικά προγράμματα. Σε πολλές χώρες. και αναγνωρίζεται η σημασία του. Ευχαριστώ. Δύο ομιλητές έχουν ζητήσει ακόμη τον λόγο. Θέλει κάποιος να θέσει ερώτημα. Μαρία Χόιμπου και ο κ. Ζέλεβεν. Η πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επανέλθουμε λίγο στο θέμα της δραστηριοποίησής σας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είπατε εισαγωγικά ότι χρηματοδοτείτε μόνο έργα που παρουσιάζουν προστιθέμενη αξία. Λογικό είναι αυτό, αφού είστε τράπεζα. Όμως, θεωρείτε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία, πρόσθετο όφελος δηλαδή, όταν ε, επενδύεται στην καταπολέμηση της φτώχειας και Υπάρχει κάποιο σχεδιασμός από την δική σας πλευρά ώστε να χρηματοδοτούνται έργα σε φτωχές χώρες στόχος των οποίων θα είναι η καταπολέμηση φτώχειας και αν ναι, τι μέτρα ελέγχου λαμβάνετε. Επίσης, άλλο ερώτημα. Εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι νομικά δεσμευτική. Εσείς έχετε ωστόσο κάποια δέσμευση να συνεργάζεστε μόνο με εταιρείες που εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επίσης, μιλήσαμε σήμερα το πρωί για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ελέγχεται προτού προβείτε σε συνεργασία με εταίρους σας αν και κατά πόσον δηλαδή έχουν επιδοθεί σε φοροδιαφυγή. Κύριε ευχαριστώ κύριε Μπέλκομ για την παρουσία σας. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού συζητήσαμε μια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που αξιολόγησε έργα που χρηματοδοτείτε εσείς στην Αφρική και μπορώ να σας πω ότι η εκτίμηση του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν εξαιρετικά θετική όσον αφορά το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των έργων που χρηματοδοτείται. Καλό θα είναι να το πούμε και αυτό εδώ ε, στην ε, Επιτροπή μας. Φυσικά δεν θα ήταν το ελεκτικό συνέδριο αν δεν είχε και κάποια σημεία ε, κριτικής. Ε, αλλά αυτά τα σημεία αφορούσαν περισσότερο την Κομισιόν και όχι την ε, τράπεζά σας. Υπόθηκε και από άλλους ότι είστε τράπεζα, το είπατε κι εσείς, και ότι χρηματοδοτείτε εν μέρη μόνο τα έργα και όχι πλήρω. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θέλετε να πάρετε και πίσω τα χρήματά σα. Και τα έργα που χρηματοδοτήσατε αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά μόνο χώρες με ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό κλίμα, κάτι που βεβαίως εξασφάλισε και εσάς, για να πάρετε πίσω τα χρήματά σα. Λογικό. Αλλά αυτό που είπε και η κυρία Χόιμπουχ είναι ότι υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο χρειάζονται και εκείνες υποστήριξη. Έχετε εσείς μηχανισμούς για την παροχή τέτοιου είδους βοήθειας σε αυτές τις χώρες. Και είπατε ότι είστε το μεγαλύτερο υπερεθνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Υπάρχουν όμως και άλλοι πιστωτές. Στη Γερμανία η Τράπεζα Ανοικοδόμησης, κάνει αυτή τη δουλειά, υπάρχουν ε, και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, υπάρχει κάποιο συντονισμός, κάποια συνεργασία με τέτοιου είδου άλλα ιδρύματα ή εσείς πηγαίνετε αυτόνομα στις χώρες ή συνεργάζεστε αυτοτελώς με τις χώρες οι οποίες απευθύνονται μόνο σε εσά, χωρίς να έρχεστε σε συνεννόηση με άλλους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, Είπατε ότι 7-8 δισεκατομμύρια είναι οι επενδύσεις σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα στοιχεία αφορούν ε, το 2013. Ένα δισεκατομμύριο πήγε στη Ρωσία. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, πώς αναλύονται τα ποσά αυτά προς την ε, Ρωσία. Έχουν ε, αλλάξει τα ποσά λόγω της αλλαγής που έχει επέλθει στη σχέση μας και στις συνθήκες που επικρατούν στη σχέση μας με την ε, Ρωσία. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ωραία, ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Βεβαίω ε, και μας ενδιαφέρουν τα έργα με προστατεμένη αξία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. και ελπίζουμε και με το IFI, το οποίο έλαβε νέα πνοή πέρυσι, για να αναλάβει και πλέον ρηψοκίνδυνα έργα σε άλλου τομεί πέραν των συνηθισμένων. Ελπίζουμε έτσι να επικεντρωθούμε περισσότερο και στην μείωση τη ανέχεια. Αυτό είναι και ο λόγο που οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτική μα επέτρεψαν ε, αυτή την ε, συμπλήρωση χρηματοδότηση. Αλλιώ δεν θα την είχαμε λάβει. Αυτό είναι το νέο σημείο εστίασης λοιπόν. Ελπίζω βεβαίως ε, αυτός ο νέος μηχανισμός, ε, αυτή η αναχρηματοδότηση είναι βέβαια ρηψοκίνδυνη. Ε, σκοπός είναι μέσω αυτών των επαναχρηματοδοτήσεων να παραμείνουμε στον τομέα ενεργή. Για το ζήτημα της φοροδιαφυγής, παρακολουθούμε με προσοχή τα όσα ε, υλοποιεί ο Δεν έχουμε ειδική ανεξάρτητη πολιτική. Αυτό εν είδη απάντηση και για το ζήτημα που αφορά τη Ρωσία. Βεβαίω και είναι θέμα συζήτηση στην τραπεζά μα. Τι θα κάνουμε με τη Ρωσία. Και πάντα υπάρχουν διλήμματα. Όμως το δίλημα για ένα δημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν είναι το πιο ουσιώδες ε, πρόβλημα γιατί αυτά τα συζητάτε εσείς εδώ, στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εάν η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης από κοινού με Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο αποφασίσει να ε, αναστείλει όλες τις επενδύσεις στη Ρωσία, τότε και εμείς θα επακούσουμε βεβαίως. και δεν θα κάνουμε κάτι στην Ρωσία. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Είμαι υπεύθυνο και για το δανεισμό στην Τουρκία. Υπήρχε παλιότερα μια τράπεζα αντέξια. η οποία, η οποία τράπεζα μπήκε σε εξυγίανση, ανασυγκρότηση, πολύ σημαντική τράπεζα δανεισμού προς την τοπική αυτοδιοίκηση και εξαγοράστηκε το 2008 ή το 2009 από τη Ρωσία. Δεν υπάρχει Ρώσος στη διοίκηση της τράπεζας, ούτε επένδυση της τράπεζας αυτής στη Ρωσία. Ουσιαστικά οι μέτοχοι άλλαξαν και ο διευθυντής της τράπεζας ήρθε απελπισμένος και είπε ισχύει ότι δεν σας επιτρέπεται πλέον να ε, συνδιαλέγεστε μαζί μας και έπρεπε να του πω ναι, δεν μα επιτρέπεται πλέον, γιατί είναι ρωσικών συμφερόντων η τράπεζα, παρότι η Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με την τράπεζα. Δεν είναι άσπρο-μαύρο τα πράγματα βέβαια, αλλά εμείς οπωσδήποτε ακολουθούμε 100% τα όσα αποφασίζονται εδώ από εσάς, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και βεβαίως προσπαθούμε να είμαστε πιο ενεργοί στην Ουκρανία και το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω η κατάσταση να σταθεροποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Και εγώ ήμουν ε, σύμβουλος χρηματοοικονομικών παλαιότερα και εγώ διάβαζα αυτές τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου με μεγάλη προσοχή και χαίρομαι πολύ που εκτιμούν τις ε, δραστηριότητές μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε βέβαια πολλά σε στενή συνεργασία. Βεβαίως και συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας ε, πάντα και θέλουμε επιχειρήσεις αυτές ε, να δρομολογούνται και με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, όμως πάντα είναι θετικό η τράπεζα να χρηματοδοτεί τι επιχειρήσει αυτές μέσω ε, κεφαλαγορών για τη χρηματοδότηση, αλλά και με την αναχρηματοδότηση, τα reflows. Πολλές φορές ε, χρηματοδοτούμε νέες επιχειρήσεις από την αναχρηματοδότηση παλαιότερων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένα πολύ οικονομικά αποδοτικό σύστημα, Πρόεδρε. Ελπίζω να τα απάντησα όλα. Αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι ήθελε να προσθέσει κάτι. Μαρία Μπάρμπαρα Τσατσνάκα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να πάρετε το λόγο στην συντομία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ε, ζήτησα πραγματικά το λόγο, αλλά ένα σύντομο σχόλιο. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ε, εισήγηση. Εκπροσωπώ την μονάδα που συντονίζει τις εργασίες ε, στο χρηματοδοτικό μέσο ACP μαζί με την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και προ το παρόν ε, καταφέραμε να έχουμε μια στενή συνεργασία στην αξιολόγηση των ε, έργων που χρηματοδοτούνται από αυτό το μηχανισμό. Ένα σχόλιο πλευρά Κομισιόν. Ποιο είναι ο στόχο ε, αυτού του IFI. Είναι να χρηματοδοτήσει ακόμα πιο υψοκίνδυνες επενδύσει. Και αυτό το στοιχείο του ρίσκου θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα, γιατί ε, το, ο μηχανισμός επενδύσεων ACP είναι ένα μέσο που έχει ως στόχο ήδη τη χρηματοδότηση σε ε, ρηψοκίνδυνα μέσα και επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προσδιορίσουμε σε αυτό το ευάλωτο ε, περιβάλλον τι μπορούμε να κάνουμε που είναι ένα ακόμα πιο ρηψοκίνδυνο ενώ ταυτόχρονα βέβαια ε, διατηρούμε όλα τα κριτήρια διαφάνειας ε, ε, και ιχνελεσιμότητας. Νομίζω ότι κάποιος άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Α, για το επόμενο θέμα. Ναι, βεβαίως και θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει. Όπως και να έχει πολύ θετική η παρέμβασή σας. σημαντικό τμήμα της ευρύτερης συζήτησης για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Ε, πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την μετατόπιση προς ε, τις μικροχρηματοδοτήσεις και βεβαίως ε, θέλουμε να μας ενημερώνετε για αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλοκόφ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Στην είσοδο της αίθουσας μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματά μας για το 2013. Και σίγουρα όταν θα είναι έτοιμα και το 2014 θα τα διαβιβάσουμε στο Κοινοβούλιο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Σίγουρα και στο μέλλον ε, θα τα ξαναπούμε. Thank you very much um, for coming here today. Uh, Thank you. Maybe see you again sometime. Thank you. Okay. Bye. Okay, Ωραία συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στο 9. Πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Ξέρετε τι συμβαίνει με το ενδιαφέρον που έχουμε για διάφορα ορυκτά. Μας μίλησε γι' αυτό και ο κύριος Ματγκέικ, τον οποίο δώσαμε βραφείο Σάχαροφ. Όπως ξέρετε η Επιτροπή μας συνέγραψε γνωμοδότηση για την καθήλια αρμόδια επιτροπή για τα ευαίσθητα αυτά ορυκτά. Από το Νοέμβριο το έχουμε συζητήσει για πρώτη φορά. Η γνωμοδότηση είναι του κυρίου Βέντα από το ΕΛΚ, ο οποίος έχει και το λόγο πρώτος και μετά θα μιλήσουν πρώτα οι σκιώδεις και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας υποβάλλω το σχέδιο γνωμοδότησής μου για το ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγών κασιτέρου, τανταλίου και Βολφραμίου, των μεταλλευμάτων του καθώς και χρυσού που προέρχονται από περιοχέ συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. όλες οι μεταφράσεις, δεν υπάρχουν ακόμη όλες οι μεταφράσεις, αλλά ελπίζω όσες έχω υπάρχουν να τις έχετε λάβει και διαβάσει. Συναντήθηκα με εταίρους μας και άλλους ενδιαφερόμενους, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προσώπους της Κομισιόν, της βιομηχανία και συναδέλφων και συναδέλφους και ο κύριος στόχος του νομοθετήματος είναι να ξεχωρίσουμε επιτέλους το θέμα της παράνομης εκμετάλλευσης ορισμένων ορικτών των λεγόμενων ορικτών, συγκρουσιακών ορικτών ή ορικτών εγκρούσεως και να το αποσυνδέσουμε επιτέλους από την εξάρτησή του για την, ε, με την ε, ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, τα ανθρωπίνα δικαιώματα, τη δημοκρατία κλπ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα συναισθηματικά, αλλά πιο λογικά, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουμε σε προτάσεις, συστάσεις για λύσεις που να είναι ρεαλιστικές και να έχουν αποτέλεσμα γιατί αφορούν και αφρικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχει τεθεί το θέμα της υποχρεωτικής πιστοποίησης, αλλά δυστυχώς όταν μερικά ορυκτά, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μερικά ορυκτά, δεν υπάρχει τρόπος εκ των υστέρων να ταυτοποιήσουμε, να δούμε από πού προέρχονται. Και επομένως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις η υποχρέωση πιστοποίηση από την άλλη μεριά θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο διοικητικό βάρος Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν γενικά ποιες είναι ακριβώς οι ζώνες συγκρούσεων, ποιο είναι, το γεωγραφικό περιεχόμενο της πρότασής μας. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΣΑΠ όπου υπάρχουν ορισμοί αυτών των περιφερειών. Αν χρησιμοποιήσουμε μόνο κατάλογο ονομάτων χωρών μπορεί να προσβληθούν να θεωρηθεί ότι στιγματίζονται και έπειτα θα πρέπει να υπάρχει και συνεχής ενημέρωση. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονό ότι μερικές χώρες υφίστανται συνεχή κρίση ή είναι σε συνεχή σύγκρουση με γείτονές τους. Ας πούμε Ουκρανία-Ρωσία. Τώρα, αν καταλάβουμε ότι πρόκειται για νέο κανονισμό θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε και αποτίμησή του, αξιολόγησή του τρία χρόνια μετά. Άρα θα χρειαστεί να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι υπερβολικά βαριά η αρχική νομοθεσία όπως έγινε με τον πρώτο κατάλογο που ξεπερνούσε την πρώτη τον πρώτο κατάλογο τριών μεταλλευμάτων και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις και για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την Ευρώπη. Κάθε ορυκτό, κάθε μέταλλο χρησιμοποιείται με ιδιαίτερο τρόπο και έχει γεωγραφικές ιδιαιτερότητες η εξόριξή του. Δεν μπορούν όλα τα ορυκτά να διακανονιστούν από έναν και μόνο νομοθέτημα ή κανονισμό. Πρώτα πρέπει βέβαια να γίνει η αξιολόγηση. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εκείνους που με βοήθησαν να συγγράψω την γνωμοδότηση αυτή, ιδίως τους Κιώδης. Αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες, ελπίζω να καταφέρουμε όλοι μαζί να πετύχουμε και συμβιβασμούς και συνδυασμούς τους. Σας θυμίζω όμως ότι αύριο οι τρεις επιτροπές, Ήλτα, Ντέβε και Άφετ, στις 2 το απόγευμα θα υποβάλουν στον ΩΣΑ αυτό το due diligence process. Ευχαριστώ κύριε Βέντα. Οι σκιώδεις τώρα, πρώτα οι σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Βάντεφο για το έργο του το θέμα αυτό. Έχει, έχουμε εκφράσει κάποιες διαφορετικές ε, απόψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα αυτών των ε, νομικών διατάξεων και το γεγονός ότι ο εισηγητής κατέληξε σε δεσμευτικό χαρακτήρα είναι κάτι που το χαιρετίζουμε και χαιρόμαστε που τα επιχειρήματά μας υπέρ αυτής της θέσης έχουν γίνει αποδεκτά ε, στην Επιτροπή και από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε από την αφετηρία ότι οι διαφορετικές δικαιοδοσίες, ιδιαίτερα σαν αφορά την Κίνα και τη ΣΥΠΑ, θα μπορούσαν να μας δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα. και πολλές φορές ενδεχομένω να μην μας έπαιρναν στα σοβαρά. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα πλέον αυτά, αυτά, τα, αυτές οι διατάξεις θα είναι υποχρεωτικές είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαφωνούμε σε ένα βαθμό ε, με, τον, κύριο, με τον εισηγητή όσον αφορά την αλυσίδα τροφοδοσίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει όλη η αλυσίδα να ελέγχεται όχι μόνο το σημείο mm. εξόριξης των μεταλλευμάτων ε, των ορυκτών και σε άλλες τομείς υπάρχουν ε, παρόμοιες διατάξεις για παράδειγμα στην ε, υγεία και την ασφάλεια όταν αν δείτε δηλαδή την παραγωγή αεροσκαφών για παράδειγμα υπάρχουν μια σειρά από απαιτήσει που ισχύουν για τα στοιχεία των ε, αεροσκαφών αυτών και πρόκειται για μια πολύ αυστηρή διαδικασία για προφανείς λόγους. Δεν υποστηρίζουμε να γίνει ακριβώς το ίδιο, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχει μια αναλογία και είναι θετική αφού το να ελέγχεται η αλυσίδα τροφοδοσίας είναι ήδη κάτι που εφαρμόζεται όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, οπότε νομίζουμε ότι θα μπορούσε να ε, επεκταθεί αυτή η πρακτική και στο θέμα που συστήματος Όσον αφορά τον, ε, το γεωγραφικό πεδίο, ε, εμείς είμαστε υπέρ του να συμπεριληφθούν και οι μελλοντικέ ζώνες συγκρούσεων, να μην υπάρχει δηλαδή ένας εξαντλητικός κατάλογος που αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουμε ότι ε, αποτελούν ε, περιοχές συγκρούσεων. Ελπίζουμε να μην αφο... Φυσικά ελπίζουμε να μην ε, επεκταθούν συγκρούσεις. Θα θέλαμε λοιπόν έναν μη εξαντλητικό κατάλογο, αλλά όχι περιγραφικό, που θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του γεωγραφικού ε, πεδίου. Όσον αφορά τον κατάλογο των ε, ορυκτών, εμείς θέλουμε να ε, επεκταθεί Φυσικά για κάθε ορυκτό θα υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την παρακολούθηση της προέλευσής τους αλλά Νομίζουμε ότι θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε και την επέκταση του καταλόγου των ορυκτών, αλλά βλέποντας τις αλλαγές θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλες όσο ε, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας ε, που αναφέρθηκε αρχικά. Είναι πολύ θετικά όλα αυτά. Θα ακούσουμε και τις απόψεις των άλλων ομάδων, αλλά νομίζω ότι υπάρχει συνένεση σε όλο το φάσμα. Αυτά είχα να πω εν γέννη από τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ. Α, έφυγε ο συνάδελφο που έχει ζητήσει το λόγο, δεν τον είδα. Λόλα Σάντσε, από πλευράς Γκουε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπήρχαν ε, πολλέ άρθμε συζητήσει ε, για αυτού ε, τους φυσικούς φόρους και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του και σε ό,τι αφορά τι τις διάφορες επιμέρους Σημαντικό είναι λοιπόν οι Ευρωπαίοι Ισογωγοί αναγνωρίζουν την κατάσταση. Για αυτό το λόγο όλα αυτά είναι πολύ ευπρόσδεκτα για μας τουλάχιστον. Και ελπίζουμε πραγματικά να τεθεί σε ισχύ και να είναι και αποτελεσματική αυτή η νομοθεσία για να αποφεύγουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, τα μεταλλεύματα που προκύπτουν από περιοχές ε, σε σύγκρουση. Θα ήθελα όμως να επισημάνω μια σειρά στοιχείων. Πρώτον, η υποχρέωση, υποχρεωτική πιστοποίηση από πλευράς ε, των επιχειρήσεων. και υποχρέωση δηλαδή της επιχείρησης να πιστοποιήσει κατά πόσο ε, έχει προέλθει αυτό το προϊόν από μια ε, περιοχή όπου υπάρχει σύγκρουση και κατά πόσο αυτά τα μεταλλεύματα πιστοποιείται ότι η εξόριξή τους δεν αποτέλεσε ε, εγγενή αιτία της πρόκλησης της σύγκρουσης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ε, μικρέ και μικρότερε επιχειρήσει, είναι σημαντική και αυτή η πτυχή. Ο ΣΑ έχει θέσει αρκετά ε, φιλόδοξου στόχου και οι, Ευρω... και ε, Είχαν πρωτοπόρο δράση σε αυτό το πεδίο. Ήρθε η ώρα λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το, την ευθύνη που ε, της αναλογεί. Αυτή ήταν η πρότασή μα. Ευχαριστώ. Τζούντις Ατζεντίνη από πλευράς Πρασίνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή για την πρότασή του και για τις τροπολογίες σου. Συμφωνώ ε, ιδιαίτερα με την αιτιολόγηση που δίνεται, δηλαδή ότι η πρόταση θα πρέπει να περάσει από την μη πρόκληση ζημίας προς ε, την, την ωφέλεια. Δηλαδή μπορεί αυτή η πρόταση να μην προκαλεί ζημία, να μην ζημιώνει, να μην βλάπτει την κατάσταση, αλλά ούτε βελτιώνει και την κατάσταση επιτόπου σε αυτές τις περιοχές ε, συγκρούσεων. Αυτό πρέπει να λέμε όχι μόνο εδώ, αλλά και στους συναδέλφους από την ΙΝΤΑ. Ο λόγος για τον οποίο αυτή η πρόταση έχει τεθεί επιτάπητος είναι ακριβώς για να σπάσει αυτή η σύνδεση μεταξύ του εμπορίου ορυκτών και της, ε, των ένοπλων συγκρούσεων. Να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Και έχω λίγο την εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει ε, να το εξετάζει ως ένα απλό εμπορικό μέτρο που δεν θα πρέπει να είναι και πολύ γραφειοκρατικό γιατί αλλιώς θα εμποδίζει το εμπόριο. Θεωρώ λαθασμένη αυτή την προσέγγιση και εξαιρετικά κοντόφθαλμη γιατί αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μακροπρόθεσμα η Ευρώπη θα προμηθεύεται τους φυσικούς ε, πόρους, τις πρώτες ύλες και ε, τα επιπλέον προϊόντα που χρειαζόμαστε στη βιομηχανία μας, πρέπει να έχουμε πολύ καλέ, μακροχρόνιες σχέσεις με τις χώρες που ακριβώς ε, έχουν τα ορυχεία που μας προμηθεύουν αυτά τα προϊόντα. Αυτή είναι η βιώσιμη προσέγγιση σε ό,τι φορά τι πρώτε ύλε. Άλλο θετικό. Ο εισηγητή προσπαθεί να εντάξει την ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει αυτά τα μέτρα σε όλη αυτή την γενικότερη προσέγγιση. Πρέπει και εμείς να το εξετάσουμε αυτό γιατί χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στη συζήτηση ως μία δικαιολογία. Μην ανησυχείτε γιατί στην πράξη θα υπάρχει αντίκτυπος επειδή θα έχουμε τα συνοδευτικά μέτρα. Ουσιαστικά όμω κανείς δεν μπορεί να μα πει ούτε τι θα είναι αυτά τα συνοδευτικά μέτρα ούτε πότε θα υλοποιηθούν και δεν μας βοηθούν αυτό να διαμορφώσουμε μία βιώσιμη βιομηχανία σε αυτές τις ε, περιοχές. Το εκτιμώ λοιπόν αυτό. Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι εξετάζεται υποχρεωτικό ε, μηχανισμό και όχι εθελοντικό. Πρέπει όμως νομίζω να διαμορφώσουμε αυτή την νομοθετική πράξη και νομίζω ότι όπως και εσείς στο μέλλον θα πρέπει να εξετάσουμε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Όχι μόνο αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις τα τρία μεταλλεύματα, παραπάνω. Για να μπορέσουμε μετά στην πορεία να τροποποιήσουμε τον κατάλογο, να προσθέσουμε νέες πρωτεσίλες. Και θα καταθέσω τροπολογίες προς αυτό τον σκοπό. Επίσης, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στην εισαγωγή πρώτων υλών ε, και προϊόντα ε, πρώτης διήλυσης, αλλά και ε, προϊόντα που έχουν ως στόχο τον τελικό καταναλωτή. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να πούνε ότι ορίστε υπήρξε ιδέως επιμέλεια και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ε, σας, να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι δεν υπήρξε καμία ζημία. Πολύ απλά γιατί οι περισσότερες οι περισσότερες συσκευές, για παράδειγμα, που αγοράζει κάποιος σε ένα ε, κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών δεν ε, κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Και τελική παρατήρηση, Πρόεδρε. Η όλη διαδικασία ε, επικεντρώνεται... Ε, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο κλάδο, όμως δεν πρέπει να μιλάμε μόνο τα ενδιάμεσα στάδια αλλά πρέπει να ε, δούμε ολόκληρη την αλυσίδα ενεφοδιασμού από την εξόρυξη μέχρι το πολυκατάστημα στην Ευρώπη. Πρέπει να το προσαρμόσουμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος μέσω της νομοθεσία, να προβλέψουμε ότι τα χιτεία εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσουν να μας ε, προμηθεύουν με τέτοια υλικά που δεν προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Και ούτε υπάρχει κίνητρο τέτοιο, γιατί η αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντελώ διαφορετική. Ακριβώ επειδή εμεί εισάγουμε τεχνολογικά προϊόντα από την Κίνα. Ελπίζω λοιπόν να σας ε, δώσω τροπολογίες που πραγματικά ε, να αναβαθμίζουν αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, Ντέιβε, θα ήθελα πραγματικά ε, να προβάλλουμε και στην ίντα ότι ο στόχος είναι η ανάπτυξη και να σπάσουμε τη σύνδεση μεταξύ των πρώτων υλών και των περιοχών συγκρούσεων. Και έτσι να λάβουμε όλες αυτές τις προτάσεις υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Κύριε κυρία... Κύριο Στέιρ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να στηρίξω κι εγώ το έργο του εισηγητή. Είναι σημαντική αυτή η αλλαγή που προτείνει, δηλαδή να περάσουμε σε υπεχρεωτική πιστοποίηση και όχι εθελοντική που προτείνει η Κομισιόν. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα σας ε, προκαλέσει έκπληξη, συνάδελφοι. Και το είπε και η κυρία Σαρχεντίνη, ότι η κυρίαρχη άποψη, ίσως όχι στην Επιτροπή, αλλά εν γέννη στο Κοινοβούλιο, είναι ότι η βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προστασία της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Από την άλλη, Υπάρχει και το άλλο επιχείρημα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η προσέγγιση λοιπόν του εισηγητή είναι ρεαλιστική Μία αλλαγή που, είναι εφικτή αυτή τη στιγμή. Να περάσουμε δηλαδή στην υποχρεωτική επιστοποίηση, διατηρώντας όμως ε, το σημείο εστίασης ε, ε, στα χιτία και σε, αυτά τα τρι, σε αυτές τις τρεις πρώτες ύλες και το χρυσό. Γνωρίζουμε τώρα και την ε, θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου, που μένως τώρα υπάρχει ο κίνδυνος. Αν πάμε πολύ παραπέρα, να μην καταλήξουμε σε καμία συμφωνία, να μην υπάρχει λοιπόν κανονισμός, το οποίο είναι πολύ χειρότερο από το να δεχθούμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, όπως προτείνει ο εισηγητής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι και ένδειξη ειλικρίνειας και από πλευρά σας θα πούμε ότι συνεχίζεται η συζήτηση και στην ομάδα μας ότι ο εισηγητής ακολούθησε μια θαραλέα αλλά και ρεαλιστική ταυτόχρονα προσέγγιση και αυτό θα πρέπει να το στηρίξουμε αν τελικά θέλουμε όχι μόνο να έχουμε μια ωραία γνωμοδότηση αλλά και μία αποτελεσματική ονοματότηση. Mr. Schofflin, maybe I mispronounce your name, you'll have to correct me. Schofflin. I think. Κύριε Σόφλεν, δεν ξέρω αν... Ε, ε, Schofflin Σόφλιν είναι το όνομά μου, αλλά το είπατε πολύ ωραία. Αλλά είναι δύσκολο για φυσικούς ομολίτες της Αγγλικής. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Παρακολούθησα με προσοχή την συζήτηση, διάβασα και τη γνωμοδότηση, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Ε, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε της ε, υποχρεωτικής ε, δηλαδή πιστοποίησης της. Ωστόσο έχω κάποιες ερωτήσεις, ελπίζω κάποιοι να μπορέσουν να τις αμβλύνουν. Γενικά είμαι υπέρ του επιχειρηματος, των επιχειρηματών που ακούσαν. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από τη θέση ότι 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ είναι παράνομο, βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο όπου ο δικός μας ε, κανονισμός θα είναι αντιπαραγωγικός. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν είναι μια κεντρική δυσκολία. Πριν από 30-40 χρόνια ένας τέτοιου είδους κανονισμός θα μπορούσε να επιβληθεί σχετικά εύκολα από την Ευρώπη. Αλλά δεν ε, είμαι βέβαιος αν τα πράγματα είναι ίδια. Και από όλα όσα έχω δει και διαβάσει υπάρχουν και κάποια δίστακτοι έμποροι που δεν συμφωνούν με τους κανονισμούς που εμείς ε, θεσπίζουμε αλλά ε, ε, θα ήταν ωραίο βεβαίως να ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο και όπως είπε και η κυρία Σαρτζεντίνη το τελικό προϊόν πρέπει να το ελέγχουμε ξέρουμε ότι υπάρχουν αδίστακτες χώρες που ε, χρησιμοποιούν σπάνιες γέες ε, και έτσι αυτά τα προϊόντα μπαίνουν στην αλυσίδα φοδοσίες μας. Υπάρχει λοιπόν κάποιος τρόπος για να θεσπιστεί κάποια υπογραφή για να ξέρουμε την ε, προέλευση του κάθε προϊόντος να μπορούμε και να μπλοκάρουμε την πώληση για παράδειγμα προϊόντων. Αυτό το κινητό για παράδειγμα να λέμε ή αυτή η τηλεόραση, αυτός ο υπολογιστής έχει κατασκευαστεί με προϊόντα από ε, παράνομης προέλευσης. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε στην ουσία μόνο τα, τα, τους μισούς μας στόχους, κάνουμε, τους μισούς μας στόχους θα μπορούσαμε να ε, ε, επιτύχουμε και ίσως ούτε καν αυτούς. Όσον αφορά την τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτού του μηχανισμού, θα έλεγα ότι ε, ένα, εθελοντικό, ένα εθελοντικό σύστημα μάλλον δεν θα ήταν αποτελεσματικό. Το είχαμε άλλωστε και πρέπει να βγάλουμε διδάγματα από αυτό. Επίσης, η αλυσίδα τροφοδοσίας είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ο ΣΑ ε, έχει αύριο μια ενημέρωση για αυτό το θέμα. Γιατί αν δεν υπάρχει έλεγχο σε όλη την έκταση τη αλυσίδας τροφοδοσία, τότε ε, κάθε ένας στην αλυσίδα τροφοδοσίας ε, θα έχει αμφιβολίες για το τι έχει συμβεί πριν από εκείνους. Υπάρχουν πάρα, πολλούς, πάρα πολλά παραδείγματα ε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει με διάφορα προϊόντα που καταλήγουν στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι και Ε, μπορεί και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή επί του θέματος αυτός. Είχαμε συζητήσει κάποτε την ε, παράνομη υλοτομία. Και όταν είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση μας για το θέμα αυτό, ήμασταν βέβαιοι ότι δεν επρόκειτο να καταλήξουμε σε συμφωνία, γιατί το Συμβούλιο θα διαφωνούσε, η Επιτροπή είχε άλλες θέσεις, αλλά στην πορεία του, του διαλόγου, 18 με 18 μήνες διέργησαν, πείσαμε το ε, Συμβούλιο. Και νομίζω ότι μπορεί να πιστεί και η Κομισιόν. Υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά μηνύματα από τον Τένις Μακουέγκε, για παράδειγμα, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη για δράση στο Κονγκό. Οι γνώμες και οι απόψεις των ανθρώπων λοιπόν αλλάζουν. Ε, οπότε ε, αυτό είναι το δίδαγμα που βγάζω εγώ δηλαδή το συμπέρασμα. Το λέω και ως ε, σοσιαλίστρια, όχι ως πρόεδρος της Επιτροπής μας, ότι μπορούμε να εξετάσουμε τέτοια ενδεχόμενα και να επιδιώξουμε να καταλήξουμε σε μια καλή λύση, όπως είπε και ο εισηγητής, ότι ο στόχος μας είναι να σταματήσουμε τη βία και τις συγκρούσεις όπως, ε, σε χώρες όπως το, η Δημοκρατία του Κονγκό και γι' αυτό δώσαμε και το βραφείο Ζαχάροφ στον άνθρωπο που το δώσαμε. Έχω Διγενική Διεύθυνση Εμπορίου και ανάπτυξη. Έχετε το λόγο, συστηθείτε κιόλας γιατί δεν ξέρω ποιος ε, είναι ποιος. Σίγνα Ράτσο, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ξεκινώ εγώ. Ευχαριστούμε για τα σχόλια. και για τη συζήτηση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα κύρια σημεία που τονίστηκαν και από τους ε, ομιλητές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι αναλογική και στοχευμένη και έχει και συμπληρωματικό χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα, στοχευμένη. Ποια, ποια είναι τα βασικά σημεία της ε, αλυσίδας τροφοδοσίας, τα χιτήρια. Ποια είναι τα χιτήρια, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, χιτήρια τα οποία είναι προβληματικά και εδώ εμπνευστήκαμε από τη δέουσα ε, επιμέλεια που προβλέπει ο μηχανισμός του ΩΣΑ αλλά η εμπειρία έχει αποδείξει από την ε, εφαρμογή των ε, νόμων μέχρι σήμερα ότι είναι αδύνατον να παρακολουθήσει κανείς την προέλευση των ορυκτών μετά το χιτήριο. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις και χώρες όπου υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ε, κλάδοι, όπου υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλυσίδες ε, τροφοδοσίας, όπως για παράδειγμα η αεροναυπηρική. Και το προβληματικό σημείο στην αλυσίδα τροφοδοσίας είναι τα χιτήρια. Γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Επίσης θέλουμε όλοι οι παραγωγοί να προέρχονται από χώρες και περιοχές χωρίς συγκρούσεις. Οι πιστοποιημένοι εισαγωγείς λοιπόν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάζουν τις, ε, τις πληροφορίες που έχουν και στους προμηθευτές τους. και αντίστοιχα κίνητρα δίνονται και για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Τώρα όσον αφορά την, ε, τον αλλαγικό χαρακτήρα της προσέγγισης που υιοθετούμε και γιατί επιλέξαμε την, την εθελοντική, τον εθελοντικό χαρακτήρα. Αφενός υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αγοράς. Ξέρετε ότι υπάρχει εταιρική κοινωνική ε, ευθύνη, υπάρχουν και οι απαιτήσει των καταναλωτών, αλλά ταυτόχρονα Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στις συγκρούσεις, ε, στις ζώνες συγκρούσεων, όπως στην Αφρική. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αυτήν την γενική προσέγγιση, όπως ο, ΣΑ. Οπότε αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν και να ε, και σε περισσότερες περιοχές. Ταυτόχρονα η δική μας προσέγγιση διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Κίνας και άλλων. Ωστόσο, γνωρίζετε ότι υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης τριών ετών στο σχέδιο κανονισμού που θα μας ε, επιτρέψει να αυξήσουμε την ε, κανονιστική ε, πίεση χωρίς όμως να προκαλέσουμε κάποιο σοκ, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ε, της ε, πιστοποίησης. Γι' αυτόν τον λόγο η εθελοντική προσέγγιση θεωρούμε εμείς ότι είναι αποτελεσματική. Μάθαμε από τη δημόσια διαβούλευση ότι οι εταιρείες ε, ενδιαφέρονται για την υπεύθυνη εξόριξη ε, Για να σας δώσω και ένα στοιχείο που το αποδεικνύει. από τις, από τις 6.000 εκθέσεις που αναμένονταν με βάση τον, ε, τον νομο, ε, μόνο 1.300 τελικά υπήρξαν και αυτό σημαίνει ότι το 20% μόνο των εταιριών μπόρεσαν να γνωρίζουν με βεβαιότητα ποια είναι η προέλευση των ορυκτών που χρησιμοποιούσαν. Γι' αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα μεταλλεύματα, τα ορυκτά που χρησιμοποιούνται στα χιτήρια. Ποια είναι η γνώμη των χιτηρίων ακόμη και λένε ότι ακόμη και με τον εθελοντικό χαρακτήρα τον θεωρούν οι, τα ίδια ως υποχρεωτικό. Γιατί αν δεν ακολουθήσουν αυτήν την ε, εθελοντική πιστοποίηση θα υποστούν αρνητικές συνέπειες, θα χάσουν τους πελάτες τους. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι η εθελοντική ε, προσέγγιση στην ουσία είναι προτιμότερη έναντι της υποχρεωτικής. Άλλη διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το γεγονός ότι ε, οι περιοχές συγκρούσεων ε, παρέχουν πολύ μικρές ποσότητες προς την παγκόσμια αγορά. Στην Αφρική είναι πιο εύκολο να καθοριστεί η υπεύθυνη εξόριξη στις περιοχές όπου που έχουμε αναφέρει. Εκεί οι εταιρείε απλώς ορίζουν σε ποιες χώρες υπάρχουν συγκρούσεις και φροντίζουν να εξορίσουν από αλλού. Αυτό είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα του Αμερικανικού νομοσχεδίου Ντόρτ Φρανκ αλλά για να βελτιωθεί η δυνατότητα των χωρών αυτών εξόρυξης, υπεύθυνης εξόρυξης. είχε δίκιο η κυρία Σαρτζεντίνη, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα διαφόρων μέτρων και πολιτικών για να αυξηθεί αυτή η δυνατότητα και φυσικά η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να το πράξει και φαίνεται αυτό από την σχετική μας ανακοίνωση και όλες οι υπηρεσίες μας το φροντίζουν ώστε μόνον οι πιστοποιημένοι πόροι να χρηματοδοτούνται και θα το λέει αυτό και στις δημοσιονομικές προοπτικές αλλά ίσως η συνάδελφός μου από την Γενική Διεύθυνση ε, εύκολα να μπορεί να σας πει περισσότερα όχι εγώ ήθελα να πω ότι όλοι οι βουλευτές εδώ έχουν περιοριστεί σε 1,5 με 2 λεπτά δηλώσεις για να πούν τα κυριότερα, τις κυριότερες ιδέες. Ε, εμάς Τώρα μας έβγαλε η Κομισιόν ολόκληρο εξάψαλμο που δεν καταλάβαμε και τα περισσότερα, όλο αριθμούς. Ε, δεν είναι τέτοια η συζήτησή μας εδώ τεχνική. Θέλουμε να ταυτίσουμε τις αδυναμίες. Αλλά δεν μου αρέσουν τέτοιου είδους κηρύγματα. Εμείς θέλουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Με συγχωρείτε. Μα οι βουλευτές είτε ελεύθεροι άμα διαφωνούν με κάτι που είπε η Κομισιόν ή θεωρούν ότι δεν είναι σωστά τα επιχειρήματά του μπορούν να το ξαναθέσουν το ερώτημά τους άμα έχουν κάτι να προσθέσουν ή αν θεωρούν ότι δεν απαντήθηκε. Αν θέλετε ξαναθέστε ερώτημα που θεωρείτε ότι δεν απαντήθηκε ή ότι είπε, ανέφερε λάθη η Κομισιόν. Πρέπει όμως τώρα να δώσουμε το λόγο Ποιο είναι ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ εδώ. Να θυμάστε και τι σα είπε η κυρία Σαρτζετίνη όμω. Ε. Ευχαριστώ. Είχα εθελοντικά πει ότι μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις, αλλά θα περιοριστώ να σας επαναλάβω ότι ήδη έχουμε αρχίσει εμείς το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό του εργαλείου συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Ανεπτυξιακού Ταμείου. Αν θέλετε και άλλες λεπτομέρειες όσο υπάρχουν βέβαια θα σας τις συμπληρώσω τις πληροφορίες που σας έδωσαν οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Βέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα καταφέρω να απαντήσω όλα τα ερωτήματα ένα προς ένα, αλλά να σας πω τα εξής. Αρχικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους, που αφορούσαν κυρίως την ε, αλυσίδα ανεφοδιασμού. Θα ξεκινήσουμε όμως από μια άλλη οπτική γωνία. Οι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ε, η καθήλυνα αρμοδιότητά μας. Ε, σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν εκπρόσωπο του ΟΣΑ που μας είπε ότι σε ορισμένες ε, αφρικανικές χώρες παρατηρείται ένα φαινόμενο της μείωσης των περιοχών ε, ακραία στόχιας. Και υπάρχει βεβαίως περιθώριο βελτίωσης ακόμα και εκεί, όμως είναι ένα πρώτο βήμα προς την εξέβρεση των απαραίτητων λύσεων. Τώρα, για αυτά τελικά προϊόντα στην ε, αλυσίδα τροφοδοσίας. Και εδώ συμφωνώ με την κυρία Σαρτζεντίνη. Κάναμε και μια συνάντηση για αυτό το στοιχείο, όμως ε, συμφωνήσαμε ότι το τελικό προϊόν Ε, ο όγκος αυτών των ορυκτών είναι αμεληταίος. Είναι τόσο μικρός, σχεδόν αμεληταίος και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο την, τον εντοπισμό της προέλευσής τους. Σε περίπτωση όμως ε, μεγαλύτερου ε, εξοπλισμού, μεγαλύτερων μηχανημάτων, όπως υπάρχει ένα αεροσκάφος, τότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Τώρα, για το γεωγραφικό πεδίο. Κάποιος ε, το ανέφερε. Υπάρχει ένας τρόπος ε, να βρούμε άλλους ε, ή να αποτέψουμε μάλλον κάποιον να βρει έναν, έναν άλλον προμηθευτή και βέβαια αυτό συνδέεται και με το θέμα της μαύρης αγοράς. Σίγουρα όπως έγινε τότε και με την ε, υλοτομία. Όλοι κατανοήσαμε ότι ε, η παράνομη ε, υλοτόμηση είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και με τα χαράς θα μπορούσα να δεχθώ συμβασμούς, όμως χάρη στη ρήτρα αναθεώρησης θα μπορούσαμε να καταθέσουμε περισσότερες τροπολογίες. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι έχει τεθεί σε ισχύ αυτός ο κανονισμός. Πρέπει να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο για να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτός ο κατάλληλος. κατά πόσο δηλαδή λειτουργεί. Συμφωνώ με την κυρία Σαντζεντίνη. ότι κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα. Ίσως θα πρέπει να μεριμνήσουμε και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συνοδευτικά μέτρα. Περιμένουμε ακόμα απάντηση σε αυτή την επιστολή που είχαν συνυπογράψει και οι σκιώδεις. Επομένω, έτσι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία συμβαστική προσέγγιση σε ό,τι φορά και τρίτη αναθεώρησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέντα. Υπερθυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Καταληκτική ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 24 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Περιμένουμε να δούμε και τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε σε μερικές εβδομάδες. Προχωράμε τώρα. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε τώρα στο σημείο 10. Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση επί του θέματο. Καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι βεβαίω η Επιτροπή Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων, ΔΡΟΑ. Η κυρία Χάουταλα είναι η συγγετριά μα ε, για τη γνωμοδότηση τη ΔΕΔΕ. Έχουν καταβληθεί τροπολογίε στην ε, έκθεσή τη και θα ψηφίσουμε απευθεία στις 5.30. Τότε θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα και να έχουν τελειώσει πιο πριν στις 5.30. Θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Ε, δεν ε, θα καταφέρουμε εξαιτία των ε, διακοπών να τα εξετάσουμε σε διαφορετικό χρόνο. Παρακαλώ όσοι θέλουν ας αποχωρήσουν ήσυχα, ιδίως εσείς εκεί στο πίσω μέρος της αίθουσας για να μην διακόψουμε την ε, συνεδρίασή μας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάουτα, πρώτα και μετά στους κοιότητες συζητητές και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω όσο περισσότερο βασίζουμε τις, ε, την πολιτική μας σε ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο πιο ε, λογικό είναι ότι θα καλούμαστε να το συνεργαστούμαστε σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την ε, ζητήματα ανάπτυξης και νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε από την πλευρά μας και ξέρω ότι ε, ο εισηγητής ε, ο κύριος Παντσέρη έχει παρόμοιες απόψεις. Όταν συνέταξα τις τροπολογίες και εξέτασα τις τροπολογίες άλλων συναδέλφων και ομάδων διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα μήνυμα προς την Κομισιόν, προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Δεν είναι ένα γενικό μήνυμα που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Έχουμε άλλες ευκαιρίες να το κάνουμε αυτό. Βλέπω όμως ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφωνίες και αυτό αντικατοπτρίζεται πλέον νομίζω και στην, ε, στο αναμενόμενο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αφού έχει υπάρξει συμφωνία επί πολλών τροπολογιών. Να αναφέρω μόνο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα των ε, δεσμευτικών κοινωνικών ρητρών στις εμπορικές συμφωνίες γενικότερα τον, τον δεσμευτικό υποχρεωτικό χαρακτήρα διατάξεων ε, σε συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας. Και υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται με, τις... Ε, ε, με ζητήματα που σχετίζονται με ε, θρησκευτικές πεπιθήσεις των ανθρώπων όσον αφορά τα... Τα... τον γενετήσιο προσανατολισμό, και τα δικαιώματα αναπαραγωγής και θέλουμε να ε, υπάρχουν αυτά ως διαστάσεις στην πολιτική μας για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Υπήρξαν κάποιες ε, τροπολογίες που κινούνταν σε άλλη κατεύθυνση. Οι προτάσεις τέλο πάντων που έλαβα, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας και να συμβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, αυτό που θέλω εγώ όμως να τονίσω είναι ότι δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υπεριαλιστικές πολιτικές αλλά να ανταποκριθούμε στην, ε, ε, στην παγκόσμια σκηνή, στην παγκόσμια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε σε βάθος τις τροπολογίες. Όσον αφορά τη συμβαστική πρόταση 2 όμως, πρέπει να πω ότι σε αυτό το θέμα και αφού μίλησα με όσους ε, πρότειναν την πρωτοβολογία 5, κύριε Μπάραιο και κύριος Βέντα, συμφωνήσαμε επί τα δική τους επιμονή ότι ακόμη και αν υιοθετηθεί η συμβαστική λύση 2 μπορούμε να, να ψηφίσουμε επί της ε, πρότασης 5. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι για τα σεξουαλικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, ε, δεν ε, προτείνω υπερψήφιση, αλλά το δεύτερο κομμάτι νομίζω ότι συμφωνεί απολύτως με όλα όσα ε, έχουμε συζητήσει. Αυτά από μένα. Αν θέλουν οι συνάδελφοι να γίνει η συζήτηση, ευχαρίστω. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 5.30 για να γίνει η ψηφοφορία. Ναι. Ε, τότε θα συζητήσουμε. Στην ημερήσια διάταξη λέει 5.30. Δεν μπορώ να τα αλλάξω τώρα, γι' αυτό λέει η Πρόεδρος αλλά έχουμε χρόνο ε, για να το συζητήσουμε ή μπορούμε να κάνουμε ένα ε, διάλειμμα για καφέ και να τελειώσουμε και να, τελειώσουμε, να επανέλθουμε στις 5.30. Έχω αγάπης ομιλητές, παρακαλώ έχετε το λόγο. Εγώ αντικαθιστώ τον Ερίκο ε, Γκερέμο που είναι ο σκιώδης μας. Ως σοσιαλιστές Θέλουμε μεγαλύτερο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Πιστεύουμε στην ανάγκη να τονιστούν τα ζητήματα πολιτισμού και περιβάλλοντος στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, πρέπει να υιοθετήσουμε ένα νομικά δεσμευτικό ε, εργαλείο ε, σε διεθνές επίπεδο που θα διασφαλίζει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτήσει βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ζώνες συγκρούσεων και σε ε, ε, περιοχές που έχουν διέλθει από συγκρούσεις ώστε να διασφαλιστεί και εκεί η, η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το ΕΛΚΟ κύριο Στήρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Χάιντι για όσα έχει κάνει. Για τη συγγραφή της γνωμοδότησης δηλαδή. Δεν μιλώ εξ ονόματός της γιατί χρειάστηκε να απουσιάσει. Αλλά ήθελα να πω ότι όπως και η συγγήτρια θεωρώ και εγώ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε πλησιάσει λίγο περισσότερο στο στόχο μας να είναι η βάση όλης της νομοθεσίας και γι' αυτό η νομοδότηση αυτή είναι αρκετά σημαντική αρκετά πιο σημαντική η Χάιντι σωστά περιέγραψε τι ισχύει ως προς τις θέσεις των ομάδων τελικά νομίζω ότι εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη γνωμοδότηση πιστεύουμε όμως ότι για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά βασίζονται τελικά στα θεμελιώδη το θεμελιωδές τώρα απ' όλα είναι το δικαίωμα στη ζωή και αυτό ήθελα να το τονίσω γιατί η ίδια διατύπωση υπάρχει και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών, στην Ευρωπαϊκή Χάρτα. Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία βέβαια θα αποφασίσει η πλειοψηφία, αλλά για το ΕΛΚ τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούμε ότι δεν πρέπει να παραλείπουν το σημαντικότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, θα σου δώσω το λόγο, ορίστε. Θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε μόλις πριν ο συνάδελφο. Α, συντομότατος, συντομότατος. Δεν ζήτησε κανείς άλλος το λόγο. Μήπως η Κομισιόν δεν βλέπω κανέναν όχι. Όχι, ε, ε, ε, όχι, όχι. Χάιντι κανένα σχόλιο. Και εγώ πολύ σύντομα. Καταρχήν για τους σοσιαλιστές. Κατά τη συζήτηση θυμάμαι τι μας είπε την περασμένη φορά η Κομισιόν. Έχω κάνει μια αλλαγή στο κείμενο, μια δική μου τροπολογία. Δηλαδή δεν μιλάω πλέον για ένα δεσμευτικό νομικά εργαλείο αλλά για δεσμευτικά εργαλεία. Αυτό είναι πολύ πιο λογικό. Γιατί όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Τζον Τράγκη πριν από μερικούς μήνες μας είπε ότι το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση είναι αυτό όπως λέει και η τροπολογία του ΕΛΚ να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη τα εθνικά τους σχέδια δράσης να τα βασίσουν στις κατευθυντήρες γραμμές του ΟΗΕ. Το άλλαξα λοιπόν και είπε αν δεν απατώμε ότι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα εργαλεία ανατομέα και νομικώς δεσμευτικά. Τώρα βέβαια συζητούμε για τα ορυκτά αλλά τέλος πάντων. πριν. Ε, έκανα αυτή την αλλαγή και κύριε Στήρ παρόλο το σεβασμό που οφείλω στις πεπιθήσεις σας όταν γράφτηκε η χάρτα και εγκρίθηκε Είμαι 100% βέβαιη ότι είχε αποσαφινιστεί ότι δεν είχε θέσει άμεσα το θέμα των αμβλώσεων. Κάποτε βέβαια πρέπει και στην Επιτροπή μας να συζητήσουμε για τον οικογενειακό σχεδιασμό και τις αμβλώσεις. Γιατί πρέπει κάποτε να συζητήσουμε το θέμα των ανασφαλών αμβλώσεων ή εκτρώσεων διεθνώς. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου γίνεται δεκτή νομικά η άμβλωση σε περίπτωση βιασμού κλπ. Μπορεί η άμβλωση να γίνει με μη σωστό τρόπο, μη υγειονομικό τρόπο. Όποτε βέβαια υπάρχει κάποια ηθική διάσταση είναι πιο δύσκολη συζήτηση αλλά θα ήθελα και Πρόεδρε κάποτε να προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε όλα τα επιχειρήματα και να δούμε τι συμβαίνει γιατί είναι σημαντικό θέμα και σχετίζεται και με άλλα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών. Ευχαριστώ. Ναι, και να συνεργηθούμε και με τις άλλες ομάδες όταν νομιμοποιήθηκε η άμβλωση στη χώρα μου είχε τεθεί αυτό το θέμα των ασφαλών αμβλώσεων. Αλλά είναι για μερικούς δύσκολο θέμα και προσωπικό και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το συζητήσουμε να, μέσω των συντονιστών μάλλον. Λοιπόν, δεν βλέπω κανένας άλλος να ζητάει το λόγο, γι' αυτό φοβάμαι συνάδελφοι ότι πρέπει να διακόψουμε μέχρι τις 5.30 και τότε θα γίνουν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ σε 35 λεπτά. Okay, colleagues. I hope... Να είστε συνάδελφοι. Ελπίζω να έχετε και τις κάρτες σας. Ας κάνουμε όμως και ένα τεστ. Γιατί έχουμε πολλές ονομαστικές πληροφορίες και θα εμφαίνονται και στα πρακτικά κτλ. Λοιπόν, δοκιμαστική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ του τσαγιού και του καφέ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε ό,τι σας κατέβει get their voting cards out. We're just testing the, the technology. Να δούμε αν δουλεύει το μηχάνημα. Το μηχάνημα testing, testing, ψηφίστε παρακαλώ. 1, 2, 3, testing. Εγώ ψήφισα αποχή. Όποιος έχει δικαίωμα ψήφου να ψηφίσει. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε, έλξε. Οι περισσότεροι ήταν υπέρ του καφέ και του τσαγιού δηλαδή, της επαναφοράς της διανομής ε, καφέ και τσαγιού στις συντεδριάσεις. Λοιπόν τώρα αρχίζει η πραγματική ψηφοφορία. Την έκθεση Χάουταλα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συζητήσαμε μόλις πριν. Συμβιβαστική ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. οι άλλες καταπίπτουν. δύο υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται καρά, εγκρίνεται μάλιστα. Όλα μετά τη συμβιβαστική δύο καταπίπτουν αυτά τα από κάτω και πρέπει χωριστά συμφωνική και ως προσθήκη μάλλον να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 5 του κυρίου Βέντα καθώς και της κυρίας Μπεθερίλ Μάριο. Το δεύτερο τμήμα που αρχίζει από το τονίζει και τα λοιπά. Ως προσθήκη όμως, υπέρ, υπέρ της προσθήκης διανατάσεως της χειρός. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επτά τα Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, χές καιίετα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, χες απορρίπτεται. Α, επαλήθευση, δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες. έλξε Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. η 10 καταπίπτει 11 11 υπέρ κατά yes. επαλήθευση άρχεται ψήφισαν όλοι λίγοι απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά yes, εγκρίνεται 20 υπέρ κατά yes, εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά ποιες επαλήθευση επαλήθευση της 21 ψηφίσατε όλοι έληξε απορρίπτεται No, Wait a minute. Falls if yes, we vote. Yeah, we're going to vote amendment 23. Um... 23. Υπέρ. Κατά. Yes. Επαλήθευση. Άρχεται για την 23. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε. Ένας παραπάνω από το ΕΛ ψήφισε. Ευχαριστούμε κύριε Ρούμπικ. Τώρα εντάξει. Εγκρίνεται. 14-10. Προφορική 1 Προφορική 1 της ηγητή υπέρ Κατά Χαίρις Εγκρίνεται 24 υπέρ κατά yes εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά yes εγκρίνεται 27 υπέρ κατά yes επαλήθευση άρχεται Ψήφισατε όλοι, έληξε, εγκρίνεται. Τώρα οι δύο. προφορική δύο. Υπέρ, υπέρ της προφορικής δύο, κατά, ποιες, απορρίπτεται. Προφορική 3 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. «28 έχει καταπέσει, 29 ε, υπέρ και ο κύριος Πρέντα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά θα επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία για την 29 έληξε απορρίπτεται όχι όμως για πολύ εντάξει 30 per Κατά. Χες. Ε, πάλι η θευσία άρχεται η ψηφοφορία για την 30. Έλξε. Ισοψηφία απορρίπτεται. Για όποιους δεν το ξέρουν. Απορρίφθηκε ήδη λοιπόν. 31 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 32 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ τα χες Είμαι Μπέφρι φρυμπάριο εδώ, εδώ να σας δω εδώ να σας δω ένα ε, στη δικιά σας λοιπόν τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά άρχεται ψηφίσατε όλες γιατί τώρα καταγράφονται. Λοιπόν, έληξε. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Χάουταλα. Okay, Ωραία. Περνάμε στο σχέδιο έκθεση για την κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση. Κύριο Γκέρενς, θα μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο αυτή η ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Ε, απορρίπτεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το 18 ανοίγει άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 όχι κατά πίπτη 20 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά επαλήθευση ψηφίζουμε για το 30 ένας ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι λήξη ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά αποχές ψηφίζουμε τροπολογία 33 ψηφίστε παρακαλώ λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 34 υπέρ μαζί με την 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 36 υπέρ κατά ψηφίζουμε για την τροπολογία 36 ψηφίστε παρακαλώ τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για το 41. Τροπολογία 41. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Χωρίς συμφορία για την τροπολογία 40. Για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ για την ε, τροπολογία 4 τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 10. Τώρα. Τέλος. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ονομαστικά για τις για τις εκθέσεις. Θα γίνει λοιπόν ψηφοφορία τώρα για το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται 21 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκέρενς, παρό το γεγονός ότι δεν βρίσκεται εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περάμε στην έκθεση απαλλαγή. Έχουμε δύο τέτοιες εκθέσεις. Η πρώτη αφορά το γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά έχουμε μια δεύτερη για το EDF. Πρώτα όμως θα ψηφίσουμε για τον Νομοδοτήσεις μάλλον και οι δύο. I'm there's been a technical problem on the... Α, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα με την ε, προηγούμενη ε, ψηφοφορία. Επιστρέφουμε λοιπόν στην έκθεση που ψηφίσαμε πριν και πάλι με ονομαστική κλίση δεν λειτουργήσε πριν το σύστημα. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, για το σχέδιο έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εντάξει τώρα. Ωραία. Ίδιο μένει το αποτέλεσμα. Αλλά τώρα έχουμε και την ονομαστική κλίση που χρειαζόμαστε από τεχνική σκοπιά για το νέο σύστημα. Λοιπόν, περνάμε τώρα στη γνωμοδότηση για την απαλλαγή του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 7 τροπολογίε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Για τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Νομίζω κρίνεται. Ναι, 14 και 10. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω και πάλι είναι η ίδια πλειοψηφία. Ας θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ψηφίσουμε λοιπόν ε, τη νομοδότηση του συνολό όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρας. 23 υπέρ, 2 κατά. Ευχαριστώ. Περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Απαλλαγή το 8 του και 10ου ε αλφα. Πολύ σύντομα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση του συνολού τη, όπω έχει τυποποιηθεί, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. 23 υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Θα επανέλθουμε αύριο στις 9 το πρωί, στη ίδια αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον.